Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fahren wir fort. Es... Αγαπητοί συναδέλφοι, ας συνεχίσουμε. Είναι 3 και 4 η ώρα. Our next, unser next... Και το επόμενο σημείο είναι το σημείο 17 στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσει με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την ε, σύναψη της συμφωνίας ΕΤΑ. Δύο ανακοινώσεις, επιτρέψτε μου. Έγινε πολύ καλή ανταλλαγή απόψε πριν από λίγο με του συναντέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει εδώ και στην δική μα συζήτηση. Ήταν νομίζω πολύ παραγωγική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Κατά δεύτερον, στις επιτροπές του Κοινοβουλίου συζητήσαμε με σωστό τρόπο την ε, συμμετοχή στις επιτροπές, ε, την τοποθέτηση τη νομικής υπηρεσίας και τελικά συμφωνήσαμε και για κάποιες ε, ημερομηνίες. Ξέρετε, αυτό κανονικά αυτό το συζητούσαμε σήμερα, ότι έχουμε μια ανταλλαγή με την νομική υπηρεσία και νομική τοποθέτηση για τα κοινά μέσα και τις 38 δηλώσεις. Δεν τα κατάφερε όμως να τα ολοκληρώσει αυτά η νομική υπηρεσία. Γι' αυτό και το αναβάλαμε το σημείο αυτό για την 5η Δεκεμβρίου, πριν από την ε, ημερομηνία αυτή θα μας υποβάλει και γραπτά η νομική υπηρεσία την γνωμοδότησή της. Κατά δεύτερον, καθυστέρησαν λίγο αλλά αποφάσισαμε, αποφάσισαν μάλλον και η Επιτροπή Περιβάλλοντος να γνωμοδοτήσει. Θα ψηφίσουμε λοιπόν μάλλον στις 5 Δεκεμβρίου προκειμένου συντονιστές να ψηφίσουμε εμείς μάλλον στην δική μας επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου. Και αυτός ο λόγος συνέπεια θα έχει ότι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προσωρινά ορίζεται για τη μήνυ Ολομέλεια στις Βρυξέλλες στις 2 Φεβρουαρίου. Αυτά εισαγωγικά. Αυτές οι παρατηρήσεις. Και τώρα λοιπόν να δούμε τι σύσταση θα μας δώσει ο εισηγητής μας για τη σύναψη της συμφωνίας ΣΕΤΑ. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον εισηγητή. Thank you, Bernd. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, συναδέλφοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καναδί μα φίλοι, όλοι όσοι βρίσκονται εδώ. Όλοι σας έχετε μπροστά σας, υποθέτω, το σχέδιο σύστασής μας σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συνολική οικονομική και εμπορική Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφετέρου. Όσον αφορά το σχέδιο σύσταση, το έχετε μπροστά σας. Μπορείτε να τη διαβάσετε, να κάνετε συστάσεις. Εγώ απλά θα προσπαθήσω να πω για άλλη μια φορά εν συντομία πράγματα που ήδη γνωρίζουμε. Ότι η ΣΕΤΑ, κατά την απόψή μου, είναι η πιο σύγχρονη και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στου διαπραγματευτέ μα και χάρη στην εντολή και χάρη και στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσει, συμπεριλαμβανομένου, θα έλεγα, του γεγονότο ότι ε, ήταν εντελώ διαφανή ο τρόπο μέχρι στιγμή με τον οποίο ε, έγινε διαπραγμάτευση για αυτή τη συμφωνία. Ο Καναδάς είναι σημαντικός ε, εμπορικός και επενδυτικός ε, στρατηγικός εταίρος. Το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους στόχους που είχαν τεθεί στη διαπραγματευτική εντολή. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται το σύστημα του διεθνούς σύστημα επίλυση διαφορών με το ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε δεν θα συμπεριληφθεί το κομμάτι ICS. Επίσης ε, ξέρετε ότι έχουμε αναβάλει την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή εμπορικής στο Κοινοβούλιο γενικότερα και έχουμε χρόνο για να γίνει και η τελική και η εξέταση από τις νομικές υπηρεσίες, νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να δοθούν κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που απομένουν. Όσον αφορά το περιεχόμενο της εμπορικής συμφωνίας, το έχουμε μελετήσει επανειλημμένως μαζί με τους ε, ενδιαφερομένους και εμείς οι ίδιοι συζητώντας όλα τα ωφέλη που θα φέρει αυτή η εμπορική συμφωνία, τα οποία μόλις ανέφερα Εν συντομία, ε, εμπόριο αγαθών, εξαιρετικά σημαντικό φυσικό, φυσικά, διότι απαλήφει σχεδόν όλους τους τελωνιακούς δασμούς, εμπόριο υπηρεσιών, πολύ σημαντικό ζήτημα, θα προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές, στις ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η συμφωνία αυτή θα δώσει και το πράσινο φως για πολυάριθμες μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής διαμαρτύρονται ότι στο μέγεθός τους ε, ε, αντιστοιχούν μόλις το 1% του εμπορίου με τον Καναδά. Ελπίζω λοιπόν αφού ολοκληρωθεί και κυρωθεί αυτή η συμφωνία να αυξηθεί το 1% γιατί αυτή η συμφωνία πρωταρχικά πρέπει να ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι όπως φοβούνται κάποιοι τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ε, επίσης δεν αποτελούν κάτι κακό. Οι δημόσιες προμήθειες, ε, εξαιρετική νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ανοίγει την αγορά με τον Καναδά, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο. Ε, πολλές δραστηριότητες, οι επιχειρήσεις μας λοιπόν θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσει για να συμμετάχουν στις δημοσίες προμήθειες των χωρών αυτών ε, οι γεωγραφικές ενδείξεις ε, χαίρουν τώρα καλύτερης προστασίας ε, και θα χαίρουν καλύτερης προστασίας αφού θα έχει συναυθεί η σύμβαση αυτή και φυσικά επενδύσεις. Δεν είναι το μεγαλύτερο, ούτε το σημαντικότερο κομμάτι επενδύσει, αλλά ήταν ένα επίμαχο κομμάτι για πολλούς από εμάς. Εγώ ο δεν τις φοβάμαι, αλλά πιστεύω ότι η συμφωνία είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για μας ε, προτείνεται ένας διαφανής αντικειμενικός τρόπος επιλογής των δικαστών. Οπότε σε εμάς αναπόκειται να εμπιστευτούμε τους δικαστές που θα επιλέγουμε για τέτοια ζητήματα σε περίπτωση που προκύψουν, αν προκύψουν. Και φυσικά έχουμε και ένα ε, όργανο ερμηνείας και επειδή ε, η συμφωνία αυτή ε, θα πρέπει να εξεταστεί και από το, Εθνικό, από το Ευρωκοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, ο κύριος Λάγκεν πριν από μισή ώρα συζητούσε με συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπότε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα έχουν δημιουργηθεί ώστε να προχωρήσουμε. Αναμένω να ακούσω τα πολύτιμα σχόλιά σας όσον αφορά το σχέδιο σύστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτος ο κύριος Νόσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να έχω μια κάπως ε, νυφάλια αντιμετώπιση για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμα τη νομική γνωμοδότηση και παραμένουν ακόμα κάποιες αμφιβολίες. Πιστεύω ότι η ΣΥΤΑ είναι μια προοδευτική συμφωνία, προοδευτικού χαρακτήρα ή τουλάχιστον περιέχει προοδευτικού χαρακτήρα στοιχεία εν γέννη, με μια συνολική αντιμετώπιση. Η ΣΥΤΑ είναι μια μεγάλη κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο και μια δήλωση αν θέλετε σε παγκόσμιο επίπεδο ότι το εμπόριο και η αηφόρος ανάπτυξη δεν είναι ασύμβατη ασύμβατα στοιχεία. Στο παρελθόν υπήρχε λιγότερο ενθουσιασμό από του Καναδού για τα θέματα του περιβάλλοντο. Αλλά το γεγονό ότι έχουμε τώρα μια συμφωνία πακέτο που να περιλαμβάνει στοιχεία για τα εργασιακά, για το περιβάλλον και έχουμε και το κεφάλαιο που καλύπτει αυτά τα θέματα αποτελεί ίσω μια πρόοδο στην ιστορία των εμπορικών συμφωνιών. Η ΣΥΤΑ απαγορεύει στι δύο πλευρέ να κάνουν ε, παρεκκλήσεις από την εργασιακή ή περιβαλλοντική τους νομοθεσία για να προωθήσουν το εμπόριο. Επομένως, δεν έχει νόημα τέτοιες ε, ανησυχίες να μπλοκάρουν αυτή τη συμφωνία. Επίσης, είναι δεσμευτικές και εφαρμόσιμες οι διατάξεις της συνθήκης βέβαια δεν εμπεριέχονται στο Γενικό Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών που περιλαμβάνει και κυρώσεις. Υπάρχει ένας πιο ήπιος μηχανισμός ε, επίλυσης διαφορών σε αυτή τη συνθήκη και ίσως είναι σωστό και εδώ η Κομισιόν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει <clears throat> ε, είναι δύσκολο να έχουμε πάντα τη Γενική Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορίου άμα χρειάζεται να εφαρμόσουμε κάποιες κυρώσεις και δεν χρειάζεται η ΣΥΤΑ γι' αυτό. Επίσης υπάρχει μια δέσμευση των δύο πλευρών να γίνει μια ε, αναθεώρηση σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να προσαρμοστούν αν χρειάζεται η διατάξη για το περιβάλλον και το εμπόριο ή τα εργασιακά και το εμπόριο και θα ήταν χρήσιμο η Κομισιόρα να μας δώσει ένα καλύτερο χρονοδιάγραμμα για το πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και για τα εργασιακά και για τα περιβαλλοντολογικά <clears throat> υπάρχει, υπάρχουν διατυπώσεις που επιβεβαιώνουν το τωρινό επίπεδο προστασίας με μια σαφή κατεύθυνση προς βελτίωση της προστασίας. Λοιπόν, δεν μειώνονται τα πρότυπα, αλλά ενισχύονται και αναβαθμίζονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, όταν έχουμε τον, τον Trump, ο οποίος διαμφισβητεί πάρα πολλά από τα επιστημονικά πορίσματα για το, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, όταν εμεί θέλουμε να κρατήσουμε μια στάση αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό ότι και η ΣΥΤΑ μα δίνει τέτοια επιχείρηματα. Τραμπισμό, ναι, τραμπισμό, έτσι το λέω, λέω. Η αρχή της ε, πρόληψης δεν επηρεάζει την αρχή της πρόληψης, της προφύλαξης της συνθήκη, η ΣΥΤΑ. Εγώ τη διάβασα προσεκτικά τη συνθήκη και σε δύο <clears throat> σημεία, χωρίς να αναφέρεται στην αρχή της πρόληψης, υπάρχει μια τέτοια διάταξη που έχει τον ίδιο χαρακτήρα, το άρθρο 23.2 για τα εργασιακά λένε οι συμβαλόμενες πλευρές ότι όταν υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι συνθήκες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα, σε τραυματισμό ή σε αρρώστιες, επαγγελματική αρρώστια, δεν θα χρησιμοποιηθεί η έλλειψη επιστημονικής, δεδομένης επιστημονικής γνώσης για να αναβληθεί η λήψη των απαραίτητων μέτρων. Και έχουμε κάτι αντίστοιχο για το περιβάλλον. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το θέμα. Ο Καναδάς έχει ήδη κυρώσει οκτώ από τις συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ακόμα και αν δεν το λέει συνθήκη, και μέχρι τον ε, Ιούλιο του 2017 ε, δεσμεύονται να τις κυρώσουν. Η ΣΥΤΑ βέβαια τους δεσμεύει να τηρήσουν το πνεύμα, όχι κατά ανάγκη το γράμμα, αυτών των ε, συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και επομένως αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται με την συμφωνία αυτή μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τα υψηλά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο. Μετά από την ΣΥΤΑ, μια οικονομία που να βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα θα προκύψει στον Καναδά. Υπάρχουν τρεις τομείς όπου μπορώ εγώ να εντοπίσω, όπου θα ευθυγραμμιστεί ο Καναδάς με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αυτό αφορά τη γεωργία, τα οχήματα, τα αυτοκίνητα και τα υφαντουργικά. Αυτή είναι τρεις τομείς. Επομένως, θα υπάρξει και η πίεση της οικονομίας πέρα από το γράμμα της συνθήκης που θα επιβάλλει με οργανικό τρόπο τα πρότυπα αυτά. Το δικαίωμα ρύθμισης αυτό διατηρείται από την συνθήκη, αλλά και έμεσα παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια προσέγγιση αρνητικού ε, καταλόγου. Υπάρχουν τώρα οι, κατα... οι τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται απόλυτα από το κεφάλαιο, από το παράτημα 2 και εκεί περιλαμβάνονται τομείς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μετατόπιση παραδείγματο για το σύστημα επίλυσης διαφορών. Δεν θα μπω <clears throat> σε λεπτομέρειες. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα για τη δική μου ομάδα και αντί να χάνουμε εξουσία έναντι των πολιτικών, παίρνει πίσω την εξουσία από τι πολιτικές άμα το συγκρίνεται με το προηγούμενο σύστημα ISDS, δηλαδή επίλυση διαφορών, τέλο η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κριτήρια περιβάλλοντο και ε, κριτήρια εργασιακού χαρακτήρα στις δημόσιε προμήθειε. Αυτό δίνει σημαντικές ε, βελτιώσει και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όπω λέει και η γνωμοδότηση τη επιτροπή απασχόληση. Επίση, σε ό,τι αφορά το πέρασμα από τα τελωνία και τι δοκιμασίε στα προϊόντα αυτά, αυτό ωφελεί πολύ περισσότερε μικρομεσαίε επιχείρησει που είχαν σε μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος να αντιμετωπίσουν συγκριτικά από ότι οι μεγάλε πολιτικές εταιρείε, για τι οποίε αυτό είναι ένα ελάχιστο κομμάτι του κόσμου. Με όλα αυτά, στο φω όλων αυτών, εγώ θα μπορέσω να παρακολουθήσω τη συζήτηση που θα έχουμε στου επόμενους μήνες. Χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι η συντηρητική πλειοψηφία των μελών των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα υποστηρίξει τη σύμφωνη αυτή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να αυτοπεριοριστούμε και κάπως. Γιατί χρονικά δεν θα καταφέρουμε να δώσουμε σε όλους το λόγο. Να είστε λοιπόν το δυνατόν συντομότεροι. Ιδάλλω θα πρέπει να αρχίσω να σα περιορίζω. Ο κύριο Κέμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και ξαναξεκινάμε. Είναι η μέρα τη μαρμότα σήμερα. Κάθε πρωί ξυπνάμε και επικοινωνούμε τη ΣΥΤΑ. Ναι, το ECR λοιπόν θα υποστηρίξει την πρόταση να δοθεί σε εγκατάσταση στην FTA. Είναι η καλύτερη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που έχει πετύχει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το μεγαλύτερο εταίριο της, ε, των ΗΠΑ, μεγάλο παράγοντας της ε, σύγχρονης οικονομίας και περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για το Ηνωμένο Βασίλειο, το θέμα των δημόσιων συμβάσεων, το γεγονό ότι ανοίγει η αγορά των δημοσίων υπηρεσιών. Ε, νομίζω ότι πάρα πολλά θετικά στοιχεία περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και όπως είπαμε ε, 99% των μη δοσμολογικών εμποδίων καταργούνται και επίσης δεν υπάρχει ελευθερία μετακίνησης ούτε πληρωμή για πρόσβαση στην αγορά αμφίδρομα. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ξαναπούμε ότι χρειάζεται ελευθερία ε, μετακίνησης ε, για να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Γιατί η ΣΥΤΑ αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Άρα συνολικά να σας πω ότι, ότι υποστηρίζω την πρόταση και να σταματήσουμε πια να ψάχνουμε εξυπνακιστικούς τρόπους να το σταματήσουμε και να το αναβάλουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επικυρωθεί το συντομότερο η συμφωνία ΣΥΤΑ. Η κυρία Σχάκε. Μαρίτσε Σχάκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα σεβαστώ και το χρονικό όριο. Αλλά Νομίζω ότι καλό θα ήταν να τα λέμε αυτά εξ αρχή για να είναι ίδια τα χρονικά όρια για όλου. Αλλά έχει δίκιο. Αυτά που είπε ο κ. Μόιζερ ήταν εύστοχα από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Οι λεπτομέρειε των όσων κάναμε τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλίσουμε ότι θα κινηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο για τα φλέγοντα θέματα της ε, ΣΕΤΑ και τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που ανοίγει αυτή η συμφωνία. Επικοδομητικός τρόπος που θα δώσει μεγάλες ευκαιρίες, θεωρώ, στους λαούς μας και είναι σαφές από το τελικό αποτέλεσμα ποια ήταν η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι περήφανη λοιπόν γι' αυτό. Εργαστήκαμε για να τονίσουμε διάφορες πτυχές τις οποίες προέβαλαν οι διάφορες πολιτικές ομάδες και καταφέραμε ευρεία πλειοψηφία γενικότερα για την υποστήριξη των ε, τροπολογιών μας. Να δούμε πώς θα αλλάζει και στα μεταξύ όμως ο κόσμος. Να μην χάνουμε χρόνο. Νομίζω ότι ο Καναδάς είναι βασικός υπερκαδικός εταίρος, πιο σημαντικό σήμερα και πριν από ένα μήνα. Σας έγκρισουμε πριν από ένα μήνα. Ένα σημαντικό σύμμαχος, ένα εταίρος με τον οποίο μοιραζόμαστε αξίες και νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε συγχρόνως σε έναν διακόσμο ταβαλέμανο κόσμο για να προσαρμοστούμε αλλά και να προσαρμόσουμε και το σύστημα εμπορικών κανόνων και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς προστασίας ε, του εμπορίου και σε ό,τι αφορά και ένα διεθνές δικαστήριο και πραγματικά στον αγώνα αυτό δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο σύμμαχο παρά τον Καναδά. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο επικυρώνουμε και προσπαθούμε να επικυρώσουμε πλευρά της Ευρώπης ε, δοκιμάζει τα όρια της υπομονής τους ε, των Καναδών. Ελπίζω πια όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και το χρονοδιάγραμμα το οποίο και πάλι έχει αλλάξει προς μεγάλη απογοήτευση της ομάδας μου να γίνει πλέον σεβαστό από όλους εδώ στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και οι τελευταίοι μήνες και όσα συνέβησαν τονίζουν ότι φυσικά πολλά έχουμε να κερδίσουμε από τη σύμφωνη αυτή, αλλά και πολλά έχουμε να χάσουμε αν δεν δράσουμε υπεύθυνα και δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα προφανώς έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ακόμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, χτες 455 ε, ευρωπαϊκές και καναδικές ε, ε, οργανώσεις προέβησαν σε δηλώσει όπου και προέταξαν τις οκτώ βασικές τους ενστάσεις σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Μιλάμε για 455 οργανώσεις οι οποίες έχουν μεγάλο, καλύπτουν μεγάλο φάσμα και έχουν διεξαγάγει σοβαρές μελέτες για τις τα Είχαν και το χρόνο άλλωστε. Και πλέον ε, υποβάλλουν σημαντικές ενστάσεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να προτείνω το εξή. Είναι πλέον ε, η σειρά του Κοινοβουλίου να αποφασίσει τι θα υποστηρίξει. Να αποφασίσουμε Ποια θα είναι η απάντησή μα στα 8 αυτά σημεία, στι 8 αυτέ προτεραιότητε και τι ενστάσει που προέβαλαν οι 455 οργανώσει. Θα ήθελα να τα αναφέρω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικά σημεία αυτά. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι οι 455 ενώσει οργανώσει με όλε τι διαφορετικέ επιχειρήσει που εκπροσωπούν αναφέρουν τα 8 αυτά παραδείγματα. Καταρχά η ΣΥΤΑ δίνει στου αλλαταπούς επενδυτές τους ε, τη δυνατότητα να καταγγείλουν και να υπονομεύσουν περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα. Υπονομεύει τις δημόσιες υπηρεσίες, ε, ισότητα φέρνει, τα, οι κανόνες για τα εργασιακά και το περιβάλλον δεν μπορούν να απαιτηθούν και καθιστά τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ευάλωτη σε οικονομική κρίση. Η ΣΥΤΑ ε, επίσης ε, υπονομεύει τη βιώσιμη γεωργία, την ιδιωτική σφαίρα και την προστασία των δεδομένων και εμποδίζει την δημόσια διαμορφώση πολιτική. Για αυτά τα πέντε σημεία λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Και θα ήθελα πραγματικά να καταλήξουμε σε μια τοποθέτηση για τα οχτώ αυτά σημεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι λοιπόν η ευθύνη μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την υπόθεση ακούω όλους όσοι υποστηρίζουν αυτή τη συμφωνία καλούμαστε στη, ενώπιον της συλλογική μας και ατομικής μας ευθύνης ενώπιον των ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, για τις ελευθερίες τους, για τις θέσεις απασχόλησης στο μέλλον, την πρόκληση που μας αναμένει με το Καναδά, τις ΗΠΑ του Τραμπ. Ενημερωτικά και μόνο, κατά τη διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση ε, αυτής της ε, συμφωνίας έγινε για να φοβήσουμε τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Ο Ομπάμα πριν τη συμφωνία του Παρίσιου είχε πει δεν θα την κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Ο Τριντό λοιπόν, ο σύγχρονος αυτός άνθρωπος, θα δείτε πώς θα ε, γίνει σύμμαχος του Τραμπ για την εξαγωγή ασφαλτούχου, ασφαλτούχου άμμου. Όταν μιλάμε λοιπόν για πολιτισμό και για ευημερία της ανθρωπότητας, σας πάρουμε το παράδειγμα του κλίματος. Δεν είναι καλή η συμφωνία αυτή για το κλίμα. Και ποια είναι η δική μας ευθύνη. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που μας παρουσίασε μια εξήγηση την οποία δεν κατάλαβα πολύ καλά. Δεν είμαι βέβαια και νομικός, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είχαν επιληθεί τα πάντα. Από τις 38 ερμηνείες, ε, ερμηνευτικές δηλώσεις, ε, ε, λάβαμε την απάντηση της ε, νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν που ήταν λίγο διαφορετική, ειδικά όσον αφορά την ικανότητα, τη δυνατότητα μια χώρα να διακόψει προσωρινά την υλοποίηση ή κάτι πιο ε, περίεργο ακόμα. Η νομική υπηρεσία της Κομισιόν ζητά από το παρόν κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια συμφωνία όπου το πιο ευαίσθητο σημείο για τα δικαστήρια διατησίας δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Τι ευθύνη λοιπόν θα δείξουμε εμείς μπροστά στους Ευρωπαίους πολίτες, πώς θα τους δείξουμε ότι ελέγχουμε ε, τη συμφωνία αυτή την οποία πρόκειται να υπογράψουμε και να κυρώσουμε ε, για το ε, επενδυτικά δικαστήρια είστε έτοιμοι να ψηφίσετε μια συμφωνία την οποία δεν γνωρίζετε εξ ολοκλήρου. Το θεωρώ πολύ παράξενο, παράδοξο. Και τι άλλη ευθύνη έχουμε πει γι' αυτό. Ακούστε τη συζήτηση που είχαμε, θυμηθείτε τη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί μαζί με την Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν υπάρχει συμπέρασμα. Δεν ξέρουμε αν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αν θα έχουμε θετικές επιπτώσεις σε κάποιους τομείς, αρνητικές σε άλλους. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Η ευθύνη μας ενώπιον του Ευρωπαίου πολίτη σήμερα, ε, δεδομένης της ανεργίας, ε, έγκυται στο να ε, συνάψουμε μια συμφωνία που θα έχει τόσο σοβαρές ε, επιπτώσεις στη γεωργία, στην απασχόληση και στις υπηρεσίες. Πρέπει να ψηφίζουμε μια συμφωνία που έχει λάβει την οριστική της μορφή και τις οποίες τις επιπτώσεις να γνωρίζουμε ε, ώστε να μην δώσουμε απλά δικαιώματα στις πολυεθνικές. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Τιτσιάνα Μπεγκίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μπω στην ουσία των διαφορών επιχειρημάτων υπέρ και κατά, όλα είναι απόψει. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πριν υπογράψει κανεί ε, ένα συμβόλαιο, δεν θα έπρεπε να το διαβάσει και να ε, ε, βεβαιωθεί ότι είναι νόμιμο, διότι την περασμένη εβδομάδα ε, απέρριψε το Κοινοβούλιο το, η προσφυγή στο δικαστήριο για τη ΣΕΤΑ με μεγάλη πλειοψηφία. Οπότε σχεδόν κανεί από εμά, τους συναδέλφους εδώ μέσα, δεν μπορεί να πει ότι δεν συμμετείχε σε αυτή την επιλογή. Και το ψήφισμα πολλών συναδελφών δεν ήταν υπέρ κατά της ε, συμφωνία, απλά ήταν ένα αίτημα ελέγχου τη νομιμότητά τη. Όπω είπε ο συνάδελφο κ. Ζαντό, θα μπορούσαμε να θέσουμε σε ισχύ ε, ένα τέτοιο κείμενο το οποίο να είναι ασύμβατο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ θα έλεγα να μην το κάνουμε, αλλά όπω φαίνεται με μειοψηφία. Εμεί λεγόμαστε Επιτροπή διεθνού Εμπορίου γιατί η δουλειά μα είναι να ελέγχουμε το διεθνέ εμπόριο και αν δεν κάνουμε αυτό τον έλεγχο γιατί να βρισκόμαστε εδώ. Η ψηφοφορία τη περασμένη εβδομάδα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αυξάνει τη δυσπιστία των πολιτών ω προ του πολιτικού και να δημιουργεί προβλήματα στη διαφάνεια λόγω τη παγκοσμιοποίηση. και δεν είναι η μόνη περίπτωση όπου αποτυγχάνει έτσι η Επιτροπή μας. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες μας δίνουν μόνο την επίσημη δυνατότητα να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε μια διεθνή συμφωνία. Αλλά η κύρωση πρέπει να συνοδεύεται από ένα ε, ψήφισμα τη Επιτροπή. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ στην ΙΝΤΑ, όχι μόνο σε επίπεδο ομάδων, να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Αλλά δεν μπορεί όλο αυτό να γίνει ανεφόρον. Το χρωστάμε στου πολίτε, ε, των οποίων την εμπιστοσύνη ζητάμε. Okay, ομιλητέ ακόμα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι και περιεκτικοί. Κ. Φιέλνερ, ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω το, αυτό το οποίο είναι αδυνατό. Να πάρω ένα ε, σουηδικό σχήμα λόγου και να το μεταφέρω στα αγγλικά. Δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν μπορείτε να δείτε το δάσος λόγω όλων αυτών των δέντρων. Α, υπάρχει αυτό. Ναι, το καταλάβατε. Μπράβο. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις συζητήσεις για τη ΣΥΤΑ εστιάζουν τόσο πολύ σε όλες τις μικρολεπτομέρειες και δεν παίρνουμε πρέφα την μεγάλη εικόνα. Ας καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτή η συμφωνία και τι προσπαθεί να επιτύχει και τι θα επιτύχει. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να συμπεράνουμε το εξή. Είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Με την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορίας αυξηθήκαν οι, εκ, οι εξαγωγές μας κατά 55% και 40% σκορές. Η ΣΥΤΑ είναι πιο πλήρη συμφωνία και γι' αυτό υπάρχουν καλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει ακόμα σε πιο καλά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση με άλλες νητικές συμφωνίες. Οι περισσότερες μειώσεις δασμών θα ξεκινήσουν από τώρα και στη γεωργία ακόμα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ πλοκά όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε εξετάσει όλα αυτά τα θέματα. Για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς, 92% των δασμών θα εξανεμιστούν. Θα έχουμε πρόσβαση σε αγορές προμηθειών 30 δισεκατομμύριων ευρώ το χρόνο. Θα έχουμε σαφείς κανόνες για την πνευματική ιδιοκτησία αυτό σημαίνει ότι οι φαρμακευτικές μας εταιρείες θα έχουν σαφή δικαιώματα στην καναδική εταιρεία, στην καναδική αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τομεί υπηρεσιών που ήταν μέχρι τώρα κλειστοί θα ανοιξούν σε ανταγωνισμό. Τηλεπικοινωνίες, ε, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια και θαλάσσιες μεταφορές. Αυτά όμως δεν είναι μονάχα πλέον εκτήματα για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά είναι επίσης και ωφέλη για τους καταναλωτές μας που θα έχουν περισσότερα προϊόντα, καλύτερα, καλύτερης ποιότητας, καλύτερα τρόφιμα, καλύτερες υπηρεσίες με τα ίδια πρότυπα προστασίας των καταναλωτών. Το να πούμε όχι <clears throat> δεν είναι μονάχα ανεύθυνο, είναι ακατανόητο. Ε, κυρία Τζούλιν τον Ντάρλινγκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελέγχθηκαν ήδη κάποια από τα πράγματα που ήθελα να πω. Εγώ πιστεύω ότι είναι θετικό ότι καθυστερεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα και την Ολομέλεια μέχρι του χρόνου, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ευρεία συζήτηση σε σχέση με τη ΣΥΤΑ και σε σχέση με τι εμπορικέ συμφωνίε σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η θέληση ήταν σαφώ σαφή σε πολλέ επιτροπέ και από πολλού βουλευτέ σε άλλε επιτροπέ. Αν δούμε την εμπειρία του ψηφίσματο, τι τύπο που ήσασταν εσεί, Πρόεδρε, ο εισηγητή, Ένα από του τρόπου για να υπάρξει μια μεγάλη διαπαραταξιακή συνένεση είναι να συμμετάσχουν στο περισσότερο περισσότεροι βουλευτέ του Κοινοβουλίου και όργανα του Κοινοβουλίου περισσότερο, ώστε να ξέρουν όλοι ότι μπόρεσαν πράγματι να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Γιατί η έλλειψη συμμετοχής είχε δημιουργήσει προβλήματα στο Κοινοβούλιο. <clears throat> Το αρνητικό στοιχείο της καθυστέρησης είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θα μπορέσω να ψηφίσω γιατί θα είμαι σε άδεια μητρότητος. Αλλά θα σας σκέφτομαι κατά τη διάρκεια των οδυνών τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και θέλω επίσης να αναφέρω κάτι άλλο το οποίο ενέχθη στη συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Καθώς είτε οι εμπορικές συμφωνίες περνάνε από τα δοσμολογικά σε θέματα προδιαγραφών και κανόνων, πρέπει να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη διαδικασία διαλόγου με τα Εθνικά μας Κοινοβούλια και η σημερινή με τα Εθνικά Κοινοβούλια ήταν πολύ ενδιαφέρουσα υπό αυτή την έποψη. Ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι σημαντικό για τη ε, διαδικασία της ΣΥΤΑ. Σας λέω, ακόμα και αν ψήφιζα εγώ θα ακολουθούσα μια γραμμή που θα επιλέξει η Εθνική μου Αντιπροσωπή. Αυτό το οποίο έγινε σαφές από τη συζήτηση του Στρασβούργου την προηγούμενη εβδομάδα για το ερμηνευτικό εργαλείο και για την δήλωση, για τα, τις 38 δηλώσεις, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτές οι δηλώσεις, αυτά τα έγγραφα έχουν αλλάξει τη γνώμη πολλών συναδέλφων γιατί ήταν σημαντικά έγγραφα είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώ θα τύχουν σεβασμού σε νομικό επίπεδο, πώ θα έχουν το ίδιο ειδικό βάρο με τη συνθήκη ενώπιον μια δικαστική ενδεχόμενη διαδικασία. και γι' αυτό θέλουμε να ξέρουμε και την άποψη τη νομική Υπηρεσία Κομισιών και του Κοινοβουλίου για το καθεστώ αυτών των εγγράφων. Πιστεύω ότι να υπάρξει πλήρη σαφήνεια μέχρι ότου φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Και αυτό είναι απαραίτητο γιατί υπάρχουν ακόμα αποκλίνουσες απόψει έξω από το Κοινοβούλιο για το αν αντιμετωπίζονται σωστά όλες οι ανησυχίες. Δεν είναι σωστό να πούμε ότι έχουν καλυφθεί και καταπλανηθεί όλες οι ανησυχίες. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμα για τη ΣΥΤΑ. Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι που εξακολουθούν να ανησυχούν και τελευταίο σημείο, πάρα πολύ σύντομα, η βελτίωση των ε, εργασιακών δικαστημάτων, δικαιωμάτων και του επενδυτικού δικαστηρίου, του παγκόσμιου δικαστηρίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς θα εμπλέκονται οι ευρωβουλευτές αν κυρωθεί η ΣΥΤΑ και υπάρξουν τέτοιες ε, ρυθμίσεις. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να εμπλακούμε στη διαδικασία εφαρμογής. Ευχαριστώ. Η Καρολίν Γκραντς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για μένα είναι ιδιαίτερη η ημέρα. Ε, έχω γενέθλια, οπότε θα υπερψηφίσω. Όχι, αστείευαμε. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να συζητηθεί αυτό επαρκώς. Και η υπηρεσία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αντιληφθήκαμε ότι κάποια στοιχεία εξακολουθούν να είναι ασαφή. Και έχει σημασία το τι θα γίνει και με το νέο αυτό α, όργανο, το δικαστικό και με τις 38 δηλώσεις και όλα αυτά φυσικά θα καθορίσουν και την απόφασή μας για το ICS τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ψηφίσαμε το ψήφισμα αυτό. Γιατί θα αποφασίσαμε να στραφούμε στο δικαστήριο. Θα υποβάλει ερώτημα το Βέλγιο. Θα δούμε κατά πόσο θα υποστηρίξουμε και κατά πόσον θα το θέσουμε αυτό το θέμα στο του ICS, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα της βιωσιμότητας είναι επίσης σημαντικό. Χωρίς σου δεν ασφαλίζεται. Δεν ασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και επίσης έχουμε και την αρνητικό κατάλογο που είναι σημαντικός γιατί αν θέλουμε να είναι εξοπλισμένοι για το μέλλον αυτής της συμφωνίας ΣΕΤΑ θα πρέπει να υπάρχουν και σε άλλες συμφωνίες τέτοιες αρνητικές ε, αρνητική κατάλογοι. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα του, της αρνητικής λίστας και για το μέλλον. Έχουμε λοιπόν εκκρεμή ζητήματα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά μέχρι τι ε, 5, τις Δεκεμβρίου θα διευκρινίσουμε κάποια τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τέλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. <clears throat> Για μένα είναι μια καλή συμφωνία σε λάθος στιγμή η ΣΥΤΑ γιατί έχει επιμολυνθεί κατά κάποιο τρόπο λόγω της κατάστασης αβεβαιότητας και φόβων που προξενούνται από την ίδια την παγκοσμιοποίηση και ιδίως μετά από τον θρίαβο του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές και των συνεπειών που μπορούν να προκύψουν. Με την εμπειρία μου εμένα και με την ανάγνωση της συμφωνίας, εγώ μπορώ να καταλήξω σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, και εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Νομίζω ότι η ερμηνευτική δήλωση <clears throat> η οποία προσετέθη ήταν θετική. Γιατί τα κεφάλαια τα οποία περισσότερο απασχολούν και ανησυχούν τους πολίτες είναι η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα του περιβάλλοντος, το δικαίωμα να υπάρχουν ρυθμίσεις και αυτά ήταν πάρα πολύ ασαφή στο αρχικό κείμενο. Και βέβαια η κοινή ερμηνευτική δήλωση διασαφηνίζει τα πράγματα αυτά. Γιατί όμως δεν έγινε αυτό από την αρχή, θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν, ώστε να αποφευθεί αυτή η αμφιβολία και οι φόβοι που γεννήθηκαν. Και δεύτερον, θα μπορούσε αυτό να προβλέπεται στο μέλλον για τις μελλοντικέ συμφωνίες. Και δεύτερη, δεύτερο συμπέρασμα που αντλώ είναι ότι πολλοί άνθρωποι στις συζητήσεις όπου εγώ βρέθηκα, οι πολίτες δεν γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται με τον Καναδά, ο, για τον, στον Καναδά. Είναι το 1,38% του παγκοσμίου μπορει ο Καναδάς μόνο. Επομένως η επίπτωση στην απασχόληση δεν θα είναι τεράστια. Το ερώτημα όμως είναι τι είδους εμπορικές συμφωνίες θέλουμε να επιτύχουμε. Κάτι ακόμα το οποίο τίθεται εν ε, αμφιβολία είναι τα θέματα των δημοσίων υπηρεσιών και της ιδιωτικοποίησής τους η, ο Καναδάς δεν έχει η, ε, δημόσια υγεία. Έχει μία δαπάνη κατά κεφαλήν που είναι το μισό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι είναι πηγαίνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όλα αυτά μου δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικός κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε και στους πολίτες όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ συμφωνώ με αυτό που ελεγχθεί από πολλούς και από την Καρολάν συγκεκριμένα σε σχέση με τις ε, συνέπειες σε σχέση με την νομική αξία των δηλώσεων. Εδώ υπάρχει ακόμα μία σύγχυση. Το είπαμε και όταν συνδεθήκαμε με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα θέματα τα οποία εγέρθησαν να διαλευκανθούν. Είναι απαραίτητο όμως να σκεφτούμε και ποιες είναι οι συνέπειες. Αν δεν κάνουμε μια καλή συμφωνία με τον Καναδά, εδώ έχουμε την πιο προθυμένη συμφωνία που μπορούμε να έχουμε, δεν θα είναι ποτέ τέλεια η συμφωνία αυτή, αλλά αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να γίνει μια συμφωνία που θα αποτελεί σημείο αναφοράς. Αν δεν την εκμεταλλευτούμε αυτήν όμως και εάν παραδοθούμε στην παραπληροφόρηση που επικρατεί σε σχέση με την ΣΕΤΑ και πούμε ουσιαστικά όχι στην εμπορική πολιτική, γιατί αυτό γίνεται από πολλούς στη χώρα μου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τη βελτίωση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέω πρώτος. Η Κομισιόν, που είναι ο κύριος διαπραγματευτής για την ΣΥΤΑ, έναντι της Ιαπωνίας και του Βιετνάμ, ο εκπρόσωπος λοιπόν της Κομισιόν. Δεν είναι εύκολο το έργο σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω σύντομα να ε, εκτίσω την ποινή μου για το ΣΥΤΑ και να αποφυλακιστώ. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν έχω να κάνω σχόλια στην παρούσα φάση. Ο κύριος μας ε, ρώτησε κατά πόσο είπα χρησιμοποίησαν ποτέ διμερείς μηχανισμούς επίλυσης διαφόρων. Εγώ δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να σας εγγυθώ ότι μπορώ να σας δώσω ακριβή απάντηση, αλλά είναι σπάνιο τα περισσότερα επίμαχα ζητήματα αντιμετωπίζονται βάσει των υποχρεώσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ε, οι χώρες ε, ε, Συνήθω στις διμερεί του συμβάσει ορίζουν κάποια πράγματα πέραν που δεν καλύπτονται από τον ΠΟΕ και σε περίπτωση που υπάρχει θέμα διαφορά προτιμούν την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ για θέματα που έχουν κάποια ρυθμιστική πτυχή συμφωνήσαμε ρητά ότι θα χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ ειδικά για ε, υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά μέτρα. Αυτό αναφέρεται ρητά στην συμφωνία. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της ε, εφαρμοσιμότητας ε, του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το εμπόριο και την εργασία να κάνω μία πρώτη παρατήρηση για αυτό και για την αναθεώρηση του ICS. Η συμφωνία είναι ολοκληρωμένη. Δεν λείπει τίποτα. Αυτό που κάναμε στο μεικτό ερμηνευτικό εργαλείο στη συμφωνία με τον Καναδά και εν μέρει στη συμφωνία με την Επιτροπή, κάτι που ε, συζητήσαμε και με τον Καναδά και πιστεύουμε θα το δει ο Καναδάς είναι η συμφωνία να περιλαμβάνει μια σειρά ρητρών αναθεώρησης και σύμφωνα με τη συμφωνία δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση αυτών των ρητρών και τι αποτέλεσμα θα πρέπει να επιτυγχάνουν. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί να συμπεριλάβουμε αυτές τις ρήτρες και να πραγματοποιήσουμε την αναθεώρηση του συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα μπορεί να συμβεί μόνο αφού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Αλλιώ πέφτουμε σε επαναδιαπραγμάτευση τη συμφωνία, το οποίο έχει απορρίψει ρητά ο Καναδά και που η Κομισιόν δεν θα συνιστούσε. Η συμφωνία λοιπόν έχει ολοκληρωθεί. Θα κάνουμε αλλαγέ στη συμφωνία ω αποτέλεσμα των μελλοντικών αναθεωρήσεων προβλέπει μηχανισμό προσαρμογής της αλλαγές στη συμφωνία. Τώρα για τα ζητήματα των εργατικών ε, της βιώσιμης ανάπτυξης και ε, της βιωσιμότητας εξαρτάται, όλα εξαρτώνται από την αναθεώρηση. Αν είναι ελάχιστη ε, σημασία, θα ακολουθεί τη διαδικασία πλήρους τροποποίησης. Και εκεί θα συμμετέχει σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσει σε τροποποίηση της συμφωνίας. Ενδέχεται να χρειαστούμε και επίσημη διαπραγματευτική εντολή. Αυτό θα εξαρτηθεί από την έκταση της διερευνητικής συζήτησης με τον Καναδά επί του εκάστοτε θέματος. Για το ζήτημα του ICS, ε, του συστήματος επενδυτικών δικαστηρίων, ε, ρωτηθήκαμε κατά πόσο θα συμμετάσχει το Κοινοβούλιο σε μια τέτοια διαδικασία. Ακόμη και αν πρόκειται για μια ε, απόφαση μεκτή επιτροπή που πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο ή από το Κοινοβούλιο, είναι αδιανόητο να μην συζητηθεί εδώ το ζήτημα αυτό. Η Κομισιόν δεσμεύεται να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και να συζητά τα ζητήματα αυτά με το Κοινοβούλιο. Και πολύ ειλικρινά, για ένα ζήτημα τέτοια σπουδαιότητα και δεδομένου του ρόλου που διαδραμάτισε το Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση του νέου ICS, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Κομισιόν μπορεί να μην επιθυμεί να γίνει τέτοια συζήτηση εδώ πριν συμφωνήσει οτιδήποτε με τον Καναδά. Ε, είμαστε λοιπόν ε, πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη συμφωνία θα λάβει χώρα μόνο εφόσον υπάρχει πλήρης υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα όλων αυτών, ε, μελετάμε τώρα την ουσία. Έχουμε ξεκινήσει συζήτηση με τα κράτη-μέλη για το ICS. Τώρα ξεκινάμε τις συνομιλίες με τους Καναδούς. Οι Καναδοί ομολογοί μας, ε, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μεγάλο φόρτο εργασίες, διότι πρέπει να αλλάξουν πολλά νομοθετήματά τους για να υλοποιήσουν τη ΣΥΤΑ, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή τη στιγμή δίνουν προτεραιότητα στο νομοθετικό τους έργο. Αλλά είναι θέμα εβδομάδων για να αρχίσουμε να συζητάμε τις λεπτομέρειες ορισμένων κομματιών του ICS. Έχουμε ένα σαφές λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών. Όσον αφορά την ε, ε, θέση σε ισχύ της διάταξης για τα, για εργατικά, το ζήτημα αυτό είναι, ε, βρίσκεται υπό συζήτηση σε πολλά κράτη-μέλη και στο Συμβουλίο και εδώ. Η Κομισιόν θα χρειαστεί περισσότερη καθοδήγηση, πολιτική καθοδήγηση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το πού να κατευθύνουμε την αναθεώρηση αυτή. Και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή μελετά τι έχει συμβεί με το ζήτημα αυτό σε άλλα μέρη του κόσμου. Δυστυχώς ελάχιστα απτά αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν του, για το πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά. Αλλά το εξετάζουμε, ξανακοιτάμε μελέτες βάσει των οποίων ε, εμείς διαμορφώσαμε τη σημερινή πολιτική για την ε, εφαρμογή της αηφόρων των περιφερειών και θα έρθουμε σε επαφή με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μόλις μπορούμε. Ε, λοιπόν που δεν μπορώ να είμαι πιο ακριβής επί του θέματος αυτού, αλλά εδώ μιλάμε για μια σαφή καθοδήγηση όσον αφορά το στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, την αποτελεσματική ε, υλοποίηση, αλλά ελάχιστα είναι τα στοιχεία που έχουμε τα οποία μπορούν να μας καθοδηγήσουν για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Αυτό προσπαθούμε να βρούμε, αλλά είναι θέμα κατεπήγοντος για την Κομισιόν. Και ένα-δύο άλλα σχόλια μικρότερης σημασία. Η ΣΥΤΑ. Θέλω να είμαι απολύτω σαφή. Η ΣΥΤΑ δεν επιτρέπει σε έναν ξένο επενδυτή σε οποιονδήποτε άλλο να παρακάψει την Ευρωπαϊκή Κλιματική Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, συγγνώμη, οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Ούτε επηρεάζει τη δική μας δυνατότητα να ε, δημιουργούμε, να ρυθμίζουμε και να οργανώνουμε και να χρηματοδοτούμε τις δημόσιες ε, υπηρεσίες με τον τρόπο που επιθυμεί κάθε χώρα. Έχουμε ζητήσει το κοινό ερμηνευτικό μέσο, ο Καναδάς συμφωνεί απόλυτα. Ο Καναδάς είναι περήφανος για τις δημόσιες υπηρεσίες του, όπως πολλά από τα κράτη-μέλη μας ε, και συμφώνησε απόλυτα σε αυτό. Ε, ρωτηθήκαμε γιατί δεν τα κάναμε αυτά έτσι από την αρχή, διότι δεν σκεφτήκαμε ότι κάποια πράγματα δεν ήταν αρκετά σαφή, ίσως θα έπρεπε να το ξέραμε, αλλά τώρα που το γνωρίζουμε ότι για κάποια ζητήματα ε, τα πράγματα δεν είναι σαφή, η επόμενη συμφωνία θα είναι πολύ πιο σαφής για τα ζητήματα αυτά. Αλλά ήθελα να τονίσω ότι θα χρειαστούμε άλλη μια ερμηνευτική δήλωση για ένα σύνολο τελείως διαφορετικών ζητημάτων που θα είναι ασαφή. Δεδομένης πολυπλοκότητας της συμφωνίας αυτής, είναι απίθανο να ε, επιτυχάνεται πλήρη σαφήνεια ε, και στο μέλλον. Από την άλλη, εδώ έχουμε διδαχθεί ένα μάθημα για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε πράγματα τα οποία φαίνονται στην τελική έκθεση μια συμφωνία λιγότερο σαφή από ό,τι νομίζαμε. Θα μπορούμε έτσι να παρεμβαίνουμε σε νωρίτερο στάδιο, συζητώντα νωρίτερα με του εταίρου μα Αν τώρα ε, ολοκληρώσουμε μια διαπραγμάτευση και από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, στην Κοινωνία των Πολιτών, στο Συμβούλιο, προκύψει ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο θεωρήσαμε ότι ήταν κατά τι διαπραγματεύσει, θα πρέπει να μπορούμε να παράσχουμε διευκρινήσει ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Αλλά υποψιάζομαι ότι για άλλα ζητήματα πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε γιατί ε, εμεί δεν είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε τι αλλαγέ αυτέ ε, στι επόμενε διαπραγματεύσει μα. Τώρα το θέμα του κατά πόσο το Βέλγιο για οποιονδήποτε λόγο ε, και δεδομένου και του αιτήματο των βαλονικών αρχών. Αν το Βέλγιο λοιπόν θα ζητήσει γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Καθιστηρίου, Δικαστηρίου συγγνώμη, για τη συμμόρφωση τη συμφωνία αυτή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν θα το κρίνω. Εγώ συμμετείχα σε κάποιες από αυτές τις συζητήσεις. Συναρπαστική εμπειρία, κύριε Πρόεδρε. Αλλά οι αξιωματούχοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά δεν αντιλαμβάνονται τον τρόπο που λειτουργούν τα κράτη-μέλη. Ούτε η δική μου χώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί από μέσα, γιατί ουδέποτε εργάστηκα σε εθνικό επίπεδο. Οπότε ήταν μεγάλο προνόμιο για μένα να δω πώς λειτουργεί μια χώρα εσωτερικά για όσον αφορά ευρωπαϊκά θέματα. Ένα πράγμα είναι σαφέ. Το αίτημα διατυπώθηκε σε σχέση με τις προσθήκες που θέλουμε να ε, κάνουμε στο ICS. Και ενδεχομένως έχει νόημα Αφού αλλάζουμε το ICS, η Κομισιόν είναι βέβαιη ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε κάτι ε, που δεν συμμορφώνεται με τι συνθήκε. Αλλά αφού έχει γίνει διαπραγμάτευση και συμφώνησε και ο Καναδά και το φέρνουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για έγκριση, αν ένα κράτο μέλο επιθυμεί επαλήθευση τη συμμόρφωση με τι συνθήκε, αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Η Βαλλονική κυβέρνηση ανακοίνωσε ε, στο, ότι το κοινοβούλιο τη επιθυμεί να γίνουν αυτέ οι αλλαγέ, να δει συγγνώμη αυτέ τι αλλαγέ, να τι εξετάσει πριν αποφασίσει αν θα κυρώσει ή όχι τη ΣΥΤΑ. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε να προβεί σε αυτέ τι αλλαγέ ε, και να κάνει διαπραγμάτευση έγκαιρα με τον Καναδά. Υποψιάζομαι ότι ακόμα και αν δεν το είχε ζητήσει, αν δεν το έχουν πει κάποια άλλα κοινοβούλια, κάποια άλλα κοινοβούλια μπορεί όντω να τηρήσουν ίδια στάση ή παρεμφερή στάση. Και όπω είπα, αυτέ οι αλλαγέ δεν πρόκειται να γίνουν χωρί το παρόν κοινοβούλιο να έχει γνωμοδοτήσει. Οπότε η Κομισιόν είναι πεπισμένη ότι το αποτέλεσμα ε, θα επιτευχθεί με τον σωστό τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Παυρίτης. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν, λόγο στη, έλαβαν το μέρος της συζήτησης σήμερα. Θα ελέγξουμε όλες τις προτάσεις, θα τις ε, διερευνήσουμε και θα επανέλθουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν εμπλακεί στη συζήτηση για μια ακόμα φορά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε αυτά που είπε ο κύριος διαπραγματευτής γιατί το μήνυμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Εγώ προσβλέπω στην ε, έγκαιρη κύρωση της ε, συμφωνίας αυτής, της ΣΥΤΑ, γιατί πιστεύω ακόμα ότι το περιεχόμενο και το και ο τύπο του εγγράφου, η μορφή, πρέπει να πηγαίνουν μαζί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρο. Θα ψηφίσουμε, όπως είπα, στις 24 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προθεσμία τροπολογιών στις 9 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, 9 Δεκεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίες έχουν περιορισμένο χαρακτήρα, ναι ή όχι, για ορισμένα σημεία και θα καταλήξουμε, όπως γνωρίζετε, σε ένα πολιτικό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων οπότε οι πρόσθετες ε, παρατηρήσεις θα μπορούσαν να εκφραστούν μέσω του ψηφίσματος, ώστε και να ψηφίσουμε για το περιεχόμενο και να υπάρξει η πολιτική ανάληψη θέσεως στο ψήφισμα που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Δυστυχώς πρέπει να σας εγκαταλείψω για μισή ώρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Ντέβιτ Μάρτιν να προεδρεύσει στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ κύριε Πάμπριξ. Sorry, excuse me, I have a point of order διαδικαστική παρέμβαση μόνο για διευκρίνηση, λέει ο κύριος Στάτμουθ. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο πρόεδρος για την, τον περιορισμό για τις τροπολογίες. Είναι διαδικασία, διαδικαστικό. Μπορείτε να κάνετε ένα ναι, όχι και ένα όχι ναι, λέει ο... Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Θα προσπαθήσω να καταλάβω καλύτερα, λέει ο κ. Δάκουθ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε στο ψήφισμα είναι ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει. Δεν μπορούμε να πούμε να αλλάξουμε το τάδε σημείο ή όχι. Σημείο 18. Εξωτερικές πτυχές της διαχείρισης των τελωνίων ως εργαλείου για την ε, βελτίωση του εμπορίου. Η κυρία Μπεγκίν έχει το λόγο. Της δίνω, της δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Εμπορική Πολιτική και η Τελωνιακή Ένωση είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στενά ε, συνδεδεμένες. Όλα τα εμπορεύματα από χώρες εκτός Ευρώπης πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν από ένα τελωνίο. Αλλά μόλις μπουν στην Ένωση δεν βρίσκουν σύνορα και μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα από τη μια χώρα στην άλλη. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, πολλοί φορείς ε, επισημαίνουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών τελωνίων με αποτέλεσμα ορισμένοι φορείς να αποφεύγουν να περνούν τα εμπορεύματά τους από τα πιο αργά τελωνία προτιμώντας άλλες ε, προορισμούς με όλες τις απώλειες που αυτό σημαίνει για καταναλωτές και εργαζομένους σε κόστος και σε εργασία. Αυτό επηρεάζει το σύνολο της εμπορικής μας πολιτικής. Αυτό συμβαίνει όταν η ελέγχη είναι αυστηρότερη σε μια χώρα σε σχέση με μια άλλη. Τα παραποιημένα ή τα μη συμμορφούμενα εμπορεύματα μπαίνουν στην Ευρώπη από το πιο χαλαρό τελωνίο με συνέπεια απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων ε, και ε, εσόδων για τα τελωνία που λειτουργούν σωστά. Αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Πέντε, ξέρετε, εμπορεύματα στα 100 στην Ευρώπη είναι παραποιημένα. Και το σύνολο των παραβιάσεων βρίσκεται σε σταδιακή αύξηση ε, από το 2008 έχει διπλασιαστεί ε, μέχρι το 2015 ο αριθμός των παραποιημένων εμπορευματών από την Κίνα, το Χονγκ τα, ε, η Λευκορωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Ινδία και άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τις διμερείς τελωνιακές συμφωνίες ε, για να ενισχύσουμε την κυκλοφορία των ε, αγαθών ε, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ. Τα τελωνία πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν μέσω τελωνιακών ελέγχων την αύξηση του αριθμού ε, εμπορευμάτων που παραβιάζουν τη διανοητική ιδιοκτησία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι τα προϊόντα αυτά και αυτές οι υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 90% των εξαγωγών στην Ευρώπη, δημιουργούν το 39% των θέσεων εργασίας και μόνο το 9% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ε, πραγματοποιεί προσφυγές για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας λόγω κόστους. Η σταθερή εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων που θα έπρεπε να είναι τα ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επηρεάζει ε, την εμπορική μας πολιτική και αυτό ερεύνησα ποιες είναι οι επιπτώσεις των φαινομένων αυτών στην παραγωγή, στις επενδύσεις και στην ακυρότητα της αγοράς, ποιες επιπτώσεις έχει στα δημόσια οικονομικά και τι συνέπειες έχει στην απασχόληση για όλες τις κατηγορίες Ευρωπαίων εργαζομένων ε, που ασχολούνται με το εμπόριο και τα τελωνία. Όπως ξέρετε όσα εκτίμησε ότι μια πλήρης μεταρρύθμιση της διευκόλυνσης των συναλλαγών θα μπορούσε να μειώσει το εμπορικό κόστος έως και 10% σε παγκόσμιο επίπεδο μια μείωση έστω και 1% των εμπορικού κόστους αυξάνει το παγκόσμιο εισόδημα κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έγγραφα που σας παρουσιάζω σήμερα σας δείχνει την οδό που θέλω να ακολουθήσω ως και ήθελα να έχω τη μέγιστη συμμετοχή από σας συναδελφοί είναι κάποιε επισκέψει σε βασικά λιμάνια στην Ευρώπη και στην Ιταλία για να συναντήσουμε αρμοδίου, τελωνιακού, ε, αποστολή, ε, μεταφορείς, ε, υπευθύνου ελέγχων υγειονομικών και φυτογειονομικών και από αυτέ τι συναντήσει προκύπτει και η βάση τη εκθεσή μου μαζί με τη δική σα πολύτιμη συμβολή. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και θα παρακολουθήσω με προσοχή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στους σκιώδες να περάσουμε. Στον κύριο να από το ΕΛΚ να δώσουμε το λόγο πρώτα. Εκτός μικροφώνου. We welcome. Καλώς ορίζουμε το έγγραφο εργασία, αλλά προσβλέπουμε επίσης σε μια πιο συγκεκριμένη οριστική διατύπωση. Η τελωνιακή ένωση μεταξύ των 28 κρατών μελών θα ωφελήσει όλους. Και αυτό διδραματίζει σημαντικό ρόλο λόγω των ε, μεγάλων όγκων εμπορίου α, της Ελληνικής Ένωσης τότε που δημιουργήθηκε. Υπάρχουν διάφορα εμπορικά, μάλλον διάφορα ε, εμπόδια προς ε, το εμπόριο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και έχουμε και προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τη διοίκηση. Έχουμε περίπλοκου ε, κανόνε ε, για του πελάτε και αυτό αποτελεί, όπω σα είπα, τέτοιο εμπόδιο προ το εμπόριο. Έχουμε θέματα με την συλλογή των φόρων, οργανωμένο έγκλαμα όλο και πιο πολλά, πολλά ε, προϊόντα ελληνικού εμπορίου Έχουμε θέματα δικαιωμάτων πραγματικής ιδιοκτησίας. σε ύψος 250 εκατομμυρίων ευρώ πέρσι. Χρειάζονται μερές αντικτύπου, χρειάζονται έρευνε για να τα υπολογίσουμε όλα αυτά. Για τις ε, νέου αυτού κανόνε σε σχέση με την νομοθεσία στις Βρυξέλλες. Έχουμε λοιπόν διαδικασίες οι οποίες έχουν οριστεί πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και η βασική κριτική είναι ότι το πρόγραμμα εργασίας δεν έχει περάσει από μελέτη αντικτύπου και έχουμε διάφορα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και να μην ξεχνάμε ότι σκοπός είναι η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόληση. Θέλουμε απλοποίηση για τις μικρομεσαίες και για τις αρχές για να μειωθεί ο... η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες. Έχουμε υποχρέωση σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που παίρνουν τα σύνορα. συμφωνείτε αυτός, μπλοκάρονται στο Συμβούλιο. Και για παράδειγμα, προτεραιότητα δική μας θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα τελικά να συνάδει με το. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. κυρία Ροντρίγκας έχει το λόγο για του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό, την εισηγήθεια για το εξαιρετικό έργο και το έγγραφο εργασία που μας έφερε. Και φυσικά πάντα θα έχει τη συνεργασία και τις απόψεις μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή όσο, όσο δυνατόν. Είναι απαραίτητη η έκθεση αυτή. Θέλω να σας πενθυμίσω ότι η Τελωνιακή Ένωση είναι ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πλήρη εναρμονισμένη Τελωνιακή Ένωση. Πόρο απέχουμε παρασάγκας Έχουμε μια ενή αγορά όπου οι κανόνες και η τήρηση των κανόνων δεν γίνονται με ισόρροπο τρόπο από όλους. Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των ε, εταιριών μας και μεταξύ και των λιμένων μας. Δεν γίνεται η πιο εποφελής μεταφορά προϊόντων σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις και τα λοιπά, αλλά πηγαίνουν τα προϊόντα στους λιμένες οι οποίοι είναι πιο χαλαροί σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων και τον έλεγχο των προϊόντων. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό έχει και ε, μεγάλη επίπτωση η εφαρμογή των κανόνων και των κυρώσεων. Όλοι ψάχνουν τα λιμάνια που είναι πιο μικρά και έχουν μικρότερες κυρώσεις. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα θέμα του ανταγωνισμό σε εσωτερικό αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο. Πάντα θέλουμε το εμπόριο να είναι ένα εργαλείο όπου θα αντανακλώνται και οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ είναι κεφαλαιώδης η προστασία των καταναλωτών. Αν επιτρέπουμε να μπαίνουν προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες και τα πρότυπα. Λόγω έλλειψης κοινών ελέγχων και προτύπων ελέγχων και προδιαγραφών, τότε δεν τηρούμε αυτή την αρχή προστασία του καταναλωτή. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το να εισαχθεί ο τελωνιακό κώδικα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να απλοποιηθούν και να εναρμονιστούν οι διαδικασίε, αλλά αυτό δεν είναι το τέλο τη πορεία, δεν είναι επαρκέ από μόνο του. Κάτι άλλο σημείο που πρέπει να αναφέρουμε. Και όταν πήγαμε στο λιμένα της Βαλένθια ως αντιπροσωπεία της ΣΥΝΤΑ, είδαμε ποια είναι η πραγματικότητα των λιμανιών εκεί. Λοιπόν, πρέπει να μπορέσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε και τις αρμοδιότητες μας στον τομέα των λιμενών, των λιμένων και να κάνουμε μια σαφή έκκληση ώστε αυτή η πηγή μη προστασίας και του ανταγωνισμού να σταματήσει να υπάρχει. Οι λιμένες δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Ο Κύριο Δάρκμουθ, όχι, δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο του Ίσια. Η κυρία Σάρνε από του Φιλελεύθερου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω ότι η έκθεση η οποία μα παρουσιάζεται σήμερα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και εγώ συμμερίζομαι αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Είναι γεγονό ότι υπάρχουν τεράστιε ανισομέρειε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του τελωνιακού κώδικα και του ελέγχου τη εφαρμογή του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει να συνεχίζεται πάντα, υπάρχουν ανισομέρειε για την εφαρμογή, για τον έλεγχο. Δεν έχουμε μια πραγματική λοιπόν και αποτελεσματική τελωνιακή ένωση, ενώ πρέπει να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε, να προστατεύσουμε την ε, πνευματική ιδιοκτησία, να αναχαιτήσουμε τα παραποιημένα προϊόντα, να ελέγξουμε την ε, γεωγραφική προέλευση των προϊόντων. Ναι, χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση, χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των τελωνίων και των κρατών μελών για να μην υπάρχουν <clears throat> όλες αυτές οι ανισομέρειες και χρειάζεται και ένας αγώνας, ένα σχέδιο αγώνα κατά των παραποιημένων <clears throat> προϊόντων με κοινά πρόστιμα και κυρώσεις και ένας διάλογος σε βάθος, μια συνεργασία με τις χώρες που ξέρουμε ότι είναι παραγωγή και εξαγωγής παραποιημένων προϊόντων. Τις ξέρουμε και ίσως με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πιο ευφυή συνεργασία μαζί τους. Τέλος, <clears throat> Πιστεύω ότι με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης θα μπορούσαμε να θέσουμε και το ερώτημα για τα κράτη-μέλη της Τελωνιακής Ένωσης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είδου σχέση θέλουμε να έχουμε σε μακροχρόνιο επίπεδο με τις χώρες αυτές. Σκέφτομαι παραδείγματος χάρη την Τουρκία. Πώς βλέπουμε λοιπόν τη σχέση μας με την Τουρκία και τις πολιτικές μας σχέσεις. Ούτως ή άλλως είναι ένα καυτό θέμα, ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα και για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο διάστημα πρέπει να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους ε, της ΚΟΕ, η κυρία Μινά... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να πω δύο-τρία πραγματάκια στη συζήτηση η ίση όρια ανταγωνισμού για όλου του λιμένε στην Ένωση ασφαλώ είναι κάτι το ευκταίο. Αλλά να προσέξουμε, μην το παρακάνουμε. Και τελικά καταλήξουμε να επιβαρύνουμε του λιμένε με μεγάλο γραφειοκρατικό άχθο. Να καλέσω τον εισηγητή να αφήσει του λιμένε να υποβάλλονται και στι προτάσει για την καταπολέμηση του παρανομού εμπορίου και του εργοδότε ασφαλώ, αλλά και του εργαζόμενου. Ελπίζω η κυρία Μπεκίν επίσης να λάβει υπόψη τις διεθνείς αλυσίδες ε, προμήθειας. Και τέλος, ελπίζω ο ρόλος και του ανθρώπου αλλά και του περιβάλλοντος κυρίως να παραμείνει στο επίκεντρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος και δεν βλέπω κανένα από, τον πράσινο, από τους πράσινους και από το ΕΝΕΦ e να ζητάει το λόγο, άρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην στον κύριο Άλμπερθ στον κύριο Εγώ εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση Trade και Taxud. Έχει συνάδελφο, θα πάρει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Σουζάνε Άικ το και είμαι από την Γενική Διεύθυνση Τάξη και ανασχολούμαι τα θέματα της σχετικής νομοθεσίας και προφανώς ε, με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Είναι ιδιαίτερα παρακολουθώ τις συζητήσεις αυτές και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με το εκπαιδευτικό αυτό έγγραφο, το οποίο αντιμετωπίζει κάποιες από τις προκλήσεις ε, των τελωνιακών στοιχείων σήμερα. Γιατί αφενός, όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο και από την άλλη να προστατευτεί η κοινωνία και να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν ίσοι όροι για τους εμπόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έγγραφο προφανώς έχει να κάνει με πολλά με πολλές πτυχές των τελωνίων να απευθυνθώ και να απαντήσω σε κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Είναι σαφές ότι η Τελωνιακή Ένωση αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και συνενώνει την εμπορική πολιτική με την κοινού δασμού και προωθεί την κοινή αγορά και είναι σαφές ότι μετά από τόσα χρόνια περίπου 30 χρόνια του παλιού τελωνιακού κώδικα γιατί είναι από τα 92 ήταν πραγματικά κατεπίγουσα ανάγκη να ενημερωθεί και να υιοθετηθεί μια νέα νομοθεσία. Ο Ευρωπαϊκός Τελωνιακός Κώδικας, όπως αναφέρθηκε. Οι ανησυχίες οι οποίες ακούστηκαν πραγματικά είναι και οι δικές μας ανησυχίες. Βρισκόμαστε λοιπόν στο ίδιο, είμαστε στο ίδιο πνεύμα. Η πλήρης εναρμόνιση η αντίστοιχη και ανάλογη εφαρμογή των τελωνιακών σε όλα τα κράτη-μέλη είναι βασική σημασία. Και αυτό είναι από του λόγου για του οποίου εγκρίθηκε ο Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Κώδικα. Θα ακούσατε για τον εξυγχρονισμένο τελωνιακό κώδικα που ήταν ο προκάτοχο και πρόκειται για αναθεώρηση λοιπόν του εξυγχρονισμένου αυτού τελωνιακού κώδικα. Προχωράμε λοιπόν και παρακάτω σε ό,τι αφορά την νομοθεσία. Ο Ευρωπαϊκός λοιπόν Τελωνιακός Κώδικας ε, αποσκοπεί στην πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασίων μέχρι το 2020, πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση, το οποίο προφανώς θα υποβοηθηθεί από συστήματα αυτή και τις ίδιες απαιτήσει ε, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που θα ισχύουν σε όλες τις χώρες. Τα ίδια δεδομένα λοιπόν θα ζητούνται από τους εμπόρους, είτε εισαγάγουν είτε εξαγάγουν προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε χώρα. Και άδειες και πιστοποίησεις για τις διαδικασίες. Αυτές θα χορηγούνται με ηλεκτρονικές διαδικασίες, με ηλεκτρονικά συστήματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι παρόμοια η προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Προσπαθήσαμε να εγκρίνουμε επίση να εγκριθεί μια νομοθεσία η οποία θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και θα υπάρχουν και τα σχετικά εργαλεία που θα είναι απαραίτητα. για να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Αυτό τονίζεται και στο έγγραφο, το οποίο διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ανησυχίες που εξέφρασαν ελήφθησαν υπόψη. Θα βρείτε πολλές πληροφορίες στο, στην ιστοσελίδα της DG Taxut και μεγάλο όγκο υλικού καθοδήγησης. Περιγράφεται λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί η νομοθεσία, βέλτιστες πρακτικές, πώς θα υλοποιηθεί όλη αυτή η νομοθεσία. Καταλαβαίνω ότι οι ανησυχίε σας υπερβαίνουν ενδεχομένω και αυτά που περιλαμβάνονται στην νομοθεσία. Γιατί ο τρενικό κώδικα θα αρχίσει να ισχύει, ξεκίνησε να ισχύει μόνο από 1η Μαου 2016 και προφανώ προσαρμόζονται σταδιακά τα πληροφορικά, πληροφορικά συστήματα. Άρα, ο πλήρης αντίκτυπος θα φανεί μόνο προς τα τέλη του 2020 όταν θα έχουν καταστεί λειτουργικά όλα τα πληροφορικά συστήματα, όλα τα συστήματα IT. Κάποιες, ε, σε κάποια συστήματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ε, την χάρτινη εκδοχή, τα έγγραφα αυτά σε χαρτί. Βαθμία λοιπόν υλοποίηση. Και αυτό χρειάζεται αν πρόκειται για συστήματα τόσο περιπλοκά όσο το προκειμένο. Και θα πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να υπάρχουν διασυνδεμένα συστήματα, τα οποία θα να προετοιμαστούν και να μην υπάρχει τελικά απόκληση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Η αναφορά στην έλλειψη ομοιογένειας των λειτουργιών αυτό ξεπερνάει προφανώ την νομοθεσία. Αντιλαμβανόμαστε και τα κράτη-μέλη επίση αντιλαμβάνονται ότι ο τελωνιακό κώδικο μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο από τι τελωνιακέ αρχέ μόνο εφόσον δρούν ω μία ενιαία αρχή και συνεργαστούν αποτελεσματικά με τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνε για άλλες και επίσης να υπάρχει σωστή και ομοιόμορφη και ομοιογενή εφαρμογή. Εκδώσαμε μαζί με τα κρατημέλη, επεξεργαστήκαμε μια ανακοίνωση για τα θέματα διαχείρισης. Θα την ε, δημοσιεύσουμε στα τέλη του χρόνου. Και ο σκοπό είναι για κάποια από τα θέματα τα οποία τονίσατε και στο έγγραφο να προτείνουμε μία, ένα κοινό όραμα για την Τελωνιακή Ένωση. Πιο ομοιογενή εφαρμογή των κανόνων για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών επιτόπου και πιο μεγάλο ρόλο για τις υπηρεσίες συντονισμού των τελωνίων ενίσχυση της μεταρρύθμισης των τελωνιακών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων ανταποκρινόμενη και στις οικονομικές τους ανάγκες. Η ανακοίνωση δε αυτή θα δέξει και θέματα τα οποία και εσά σα απασχολούν σε ό,τι αφορά το port shopping, την επιλογή του λιμένα δηλαδή ανάλογα με τι ανάγκε του καθενό. Νομίζω ότι η νομοθεσία καθιστά σαφέ ότι σε όλα τα κράτη-μέλη ισχύουν οι ίδιοι κανόνε και εμεί συνεχίζουμε το διάλογο με τα κράτη-μέλη και με τον οικονομικό κλάδο προκειμένου να εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου. Αλλά φυσικά τίθεται το θέμα του εξοπλισμού, στα σύνορα, των ικανοτήτων των κρατών μελών, όλα αυτά τα πραγματεύεται η ανακοίνωση για τα θέματα διαχείρισης και μεταξύ άλλων και το θέμα της χρηματοδότησης. Θα γίνει μελέτη δικτύπου για την προετοιμασία νέων των ε, προγραμμάτων νέα γενιά στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί προφανώ ο εξοπλισμός είναι ακριβώ, ε, αυτό αποτελεί μια ανησυχία. Άλλοι είναι καλά εξοπλισμένοι, άλλοι όχι. Και υπάρχει τελικά μια ανάγκη για οικονομική υποστήριξη. Μια άλλη από τι στρατηγικέ μα ε, εξετάζει κάποια άλλα ζητήματα και ανησυχίες και ευχαριστώ να σας δώσουμε πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση ε, της επικινδυνότητας στα τελωνία ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα και ομοιομορφία ε, στη διαχείριση σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του ενιαίου τελωνιακού κωδικά αλλά και στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλειών που συμπεριλαμβάνουν και άλλους φορείς και οργανισμούς. Εμείς οθετήσαμε μια έκθεση προόδου φέτος τον Ιούλιο μετά από δύο χρόνια διότι η στρατηγική ανέρχεται στο 2014 και θα ακολουθήσουν συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα υιοθετηθούν στο Συμβουλίο στις 6 Δεκεμβρίου και εκεί θα γίνεται έκκληση προς τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να αυξήσουν τις συνέργειες μεταξύ οργανισμών και να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία. Τα συμπεράσματα θα συνοδεύουν την επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της επίσημης έκθεσης ε, ε, προόδου δεν θα επισημαίνουν ανάγκη τροποποίηση της στρατηγικής αλλά συνέχιση των προσπαθειών και τα ζητήματα που έχουν τεθεί ε, βρίσκονται υπό εξέταση. Επίσης η έκθεση αναφέρει και την οδηγία για τις κυρώσεις για την οποία γίνονται αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα οι εργασίε και η Κομισιόν καλωσορίζει τη θέση του Κοινοβουλίου όσον, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Ήταν πολύ σαφές ότι επιθυμούστε να τονίσετε την αναγκαιότητα εναρμόνισης των κυρώσεων. Εμείς εξετάζουμε τώρα και μελετάμε τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες που έχετε προτείνει ως Κοινοβούλιο σχετικά πρόσφατα. Και ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι να συνεργαστούμε και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας. ώστε κάποια στιγμή εν τέλει να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε την οδηγία. Διότι πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να εγγυηθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν κυρώσεις και θα αντιμετωπίζουν τις παραβιάσεις με ομοιόμορφο τρόπο. Κάτι που δεν συμβαίνει δυστυχώς μέχρι στιγμές. Συγγνώμη, μπορείτε να επιτεγχύνετε λίγο και να κλείσετε γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ακούσαμε πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Είναι από τα θέματα έψη της προτεραιότητας για μας. Αποτελεί κομμάτι της συνεργασίας μας με την Κίνα, αλλά και με πολλές άλλες χώρες και σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και οι κοινέ μα ε, επιχειρήσεις που συμμετέχουν η Europol, η Interpol, η OLAF και τρίτες χώρες όλες αυτές οι συνέργειες συμβάλλουν στο να σημειώνεται πρόοδος θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερος για το έγγραφο και να επισημάνω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ε, συμβάλλουμε και είμαστε διατεθειμένοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ενδεχομένω έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την εξαντλητική αυτή παρουσίαση που μας δώσατε. Πρέπει όμως να πάμε σε μια άλλη αίθουσα συνεδριάσεων στις 5. Η κυρία Μπεκίνη για να κλείσει τη συζήτηση, άμα θέλει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί αυτού του ούτως ή άλλως εργασίας το οποίο σίγουρα θα τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανησυχίες που ακούσαμε και τις επιφυλάξεις. Ε, θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο που θα είναι έτοιμο σε λίγες μέρες. Όσον αφορά αυτό που είπε η συνάδελφος κυρία Μινέρ, ήθελα να σχολιάσω την παρατήρησή σας, να επισημάνω ότι πράγματι ήδη συναντάμε, το έχουμε κάνει και ως Επιτροπή, είναι τα ορισμένους λιμενικούς φορείς ε, συναντάμε, όπως κάναμε και στην τελευταία αποστολή στη Βαλένθια τον Οκτώβριο ήταν παροντές και άλλοι ε, συναδέλφοι μεταξύ των οποίων και είμαι. Και εγώ βεβαίω, παρομοίω προσωπικά έχω συναντήσει διάφορους ε, ε, λιμενικούς φορεί στη Γένοβα, στην Τεργέστη και συνεχίζω. Οι ενησυχίε των λιμενικών φορέων είναι γνωστέ. Έχουν σημειωθεί και μου στέλνουν διάφορες προτάσεις, ε, πολύ κατάλληλες μάλιστα, πολύ ευστοχές. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή της και θα τα ξαναπούμε σε μια και θα έχουμε νεότερα σε μια επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλείσαμε το σημείο αυτό. Περνάμε στο σημείο 19 που αφορά την πρόταση για μια απόφαση του Συμβουλίου για την ε, για το εμπόριο σε, όχι, σε αεροπλάνα πολιτικής αεροπορίας. Η κυρία ε, Ροντρίγκε είναι η εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για μια συμφωνία πολυμέριου, πολυμέρη συμφωνία που καλύπτει 30 χώρες σε σχέση με το εμπόριο πολιτικών αεροσκαφών. Με το, τη συμφωνία αυτή θα ε, σταματήσουν να υπάρχουν δασμοί, αλλά αυτό βέβαια δεν καλύπτει τα στρατιωτικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κίνητρα για την αγορά των οχημάτων αυτών και καλύπτει επίσης και τις δημόσιες επιδοτήσεις στον τομέα αυτό. Είναι μία πολύ τεχνικού χαρακτήρα οδηγία, ο, σημαίνει μια αλλαγή στην ονοματολογία του τελωνιακού κώδικα, όπου αναφέρονται όλα τα προϊόντα που υπόκειται στον τελωνιακό κώδικα και επομένως το θα αλλάξει το εναρμονισμένο σύστημα κωδικοποίησης των εμπορευμάτων. Το Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή Εμπορίου για τα Πολιτικά Οχήματα ενέκρινε αυτό το πρωτόκολλο για την τροποποίηση του ηχείου παρατήματος. Επειδή αυτή τώρα η αλλαγή γίνεται στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του, δεδομένου ότι είναι τεχνικού χαρακτήρα η μεταλλαγή αυτή απαιτείται και από την δική μας Επιτροπή να την υποστηρίξουμε. Ωραία λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανένα από το EPP ή από το ECR. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεσαρνέζ εκ μέρους των Σκιωδών. Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ τεχνική είναι αυτή η διάταξη. Πρόκειται για την εναρμόνιση των κανόνων για τα πολιτικά αεροσκάφη με το παγκόσμιο κώδικα του ελληνικού χαρακτήρα. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πάρα πολύ σύντομα. Ο Χέλμουτ για την Γκουέ. Θα είμαι λίγο μακροσκελέστερος, αλλά μπορώ να συμφωνήσω με την ε, παρακολούθηση αυτή. Ξέρω ότι είναι ένα τεχνικό θέμα Θέλω να επιστρέψω την προσοχή σας σε ένα άλλο πρόβλημα. Μετά από μια πρόσφατη απόφαση του ΠΟΕ για τη διαμάχη Airbus με Boeing, θυμόσαστε ότι εφέτος ο ΙΚΑΟ συμφώνησε τα λεγόμενα μέτρα παγκόσμιας αγοράς για να μπορέσουν να ρυθμιστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από την αεροπορία που είναι η πιο βλαπτική για το περιβάλλον μορφή μεταφορών. Και σε πολλές περιπτώσεις η, αντιμετωπίζει το γεγονός ότι πολλές φορές υπάρχουν επιδοτήσεις για τους κινητήρες και τα αεροσκάφη που στρεβλώνουν την αντιμετώπιση αυτή. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο για αυτό το τεχνικό θέμα, διότι θα μας οδηγήσει ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε και αυτή την ρήτρα σε άλλες συμφωνίες που έχουν να κάνουν με την παραγωγή οχημάτων, ώστε να βρούμε μια στρατηγική η οποία θα μπορέσει να εξισορροπήσει καλύτερα την παραγωγή και τη χρήση των αεροσκαφών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Κομισιόν, ο κύριος Μέριμ, Κομισιόν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο κι εγώ. Όπω υπόθηκε, είναι καθαρά μια τεχνική μεταφορά τη εκδοχής του 2007, της έκδοσης του 2007 του εναρμονισμένου συστήματος και ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη τη ΣΥΝΤΑ για το, για το χρόνο που αφιέρωσαν σε αυτό το αρχείο. Στη Γενέβη σημειώθηκε κάποια πρόοδο, πρέπει να ξέρετε, κάποια μέλη υπέγραψαν το πρωτόκολλο. Οπότε σα ενθαρρύνω να επιταχύνετε τις εργασίες σα ε, στο βαθμό του δυνατού. Ευχαριστώ πολύ. That... Ευχαριστούμε πολύ. Επ' αυτού λοιπόν να πούμε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι Τροπολογίες 15 Δεκεμβρίου, η υιοθέτηση στην Επιτροπή 24 Ιανουαρίου. Δεν θα είναι το πιο επιμαχό ζήτημα στις 24 Ιανουαρίου πρέπει να πω και σκοπός να εγκριθεί στην Ολομέλεια στη δεύτερη ε, Ολομέλεια του Μαρτίου. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο και περνάμε στο τελευταίο σημείο, το σημείο 20, την εκθέση για την αποστολή στη Βαλένθια και στο Αλικάντε που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο. πολύ επικοδομητική η αποστολή αυτή. Δεν μπόρεσα να συμμετάσχω, αλλά η επίσκεψη στο Αλικάντε συμπερίλαβε και μια ε, επίσκεψη στο EU όπου εξέτασαν το σύστημα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και τις δυνατότητες των χωρών ε, για βελτιώσεις ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη νέα γενιά. Στη Βαλένθια έγιναν συναντήσεις με το εμπορικό επιμελητήριο της περιοχής. Έλαβε χώρα ένα δείπνο όπου ο πρόεδρος της ο περιφερειάρχης ε, ήταν παρόν. Η Βαλένθια είναι η δεύτερη εξαγωγική περιοχή της Ισπανίας και ε, εξαγεί και ε, κάνει από το Ασία και Νότιο Μεσόγειο συζητήθηκαν οι εξελίξεις του TTIP του ΣΥΤΑ και οι διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Επίσης έγινε και μια επισκέψη στο λιμάνι της Βαλένθια που είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου σε αριθμό εμπορευματοκιβωτίων και το τέταρτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη ε, και το οποίο ζητάει ομογενή ε, τρόπο ε, τελευταίων διατυπώσεων και κυρώσεων και ζήτησε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για τα τελωνία. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο για την επίσκεψη. Απλώς το μόνο που θέλω να πω είναι ότι κρίμα που δεν ήρθες, David, και θα ήταν καλό να έχεις την ευκαιρία να μεταβαίνεις σε τέτοιες τόσο ενδιαφέρουσες αποστολές. very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια θα ξαναξεκινήσουμε στις 5 την συνεδρίαση με την κοινή μας συνεδρίαση με την Επιτροπή ε, γεωργικών υποθέσεων.